ώστε να πραγματοποιήσει ένα ποιοτικό άλμα και η βιομηχανία μας, να κρατήσει την πρωτοκαθεδρία της, να διαφυλάξει τις θέσεις εργασίας και να έχουμε καθαρές μεταφορές φιλοπεριβαλλοντικές που θα μας επιτρέψουν να ανταπεξέλθουμε στην σημαντική πρόκληση που είναι η πλήρης απαλλαγή μας από τις εκπομπές άνθρακα στους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας μας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Νίμπλερ για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε εκπρόσωπε της Κομισιόν, αγαπητοί μου συνάδελφοι. Γεγονό είναι πως οι τιμές διοξιδίου του άνθρακα για τα γεωταχή και τα φορτηγά ε, προσαρμόζονται διορκώς. Χρειαζόμαστε αυτοκίνητα που εξοικονομούν ενέργεια για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αλλά οι οριακές τιμές που προτείνονται σήμερα για το 2025 και 2030 πρέπει να είναι και υλοποιήσιμες και να έχουμε τα κατάλληλα κίνητρα Γι' αυτό χαιρέτησα την πρόταση της Κομισιόν που μιλάει για ένα στόχο 30% ε, μέχρι το 2030 έτσι ώστε να υπάρχει μια κινητικότητα σε προσιτές τιμές και να διατηρήσουμε και τις θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παγκοσμίω δεν υπάρχει άλλη ανάλογη διάταξη. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν μείνει πίσω. Είναι τεράστια η ζήτηση για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πρώτα απ' όλα βεβαίως δαιμονοποιήσαμε τον δίζελ, το οποίο όμως εκπέμπει σαφώς λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα. Και τώρα δεν έχουμε κανένα κίνητρο για τα αυτοκίνητα που μπαίνουν στην ε, Μπρίζα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά είναι λάθος, γι' αυτό θα το καταψηφίσω. Εγώ δεν θέλω να έχουμε μόνο Τέσλα στην Ευρώπη προσεχώς, αλλά και κάνα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Σας ευχαριστούμε κυρία Νίμπλερ. Περνάμε στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ τώρα. Έχουμε τρεις ομιλητές και οι τρεις είναι από το ΕΛΚ. Ο κύριος Μαριάς απουσιάζει, οπότε η κυρία Σόιντροβα θα λάβει πρώτα το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι κλιματικές αλλαγές μας κάνουν όλο και πιο ευαίσθητους σε περιβαλλοντικά ζητήματα και είναι απόλυτα δικαιολογημένο κάτι τέτοιο. Ο τομέας των μεταφορών σίγουρα συμβάλλει τα μάλα στην ρήπανση την ατμοσφαιρική και επιδεινώνει και τις κλιματικές αλλαγές. Προσοχή όμως, δεν θα πρέπει ε, να κυνηγάμε ανεύθυνα τα όρια εκπομπών. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ο κύριο παραγωγό διοξιδίου του άνθρακα. Λιγότερο από 10% των εκπομπών παγκοσμίω προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, η αυτοκινητοβιομηχανία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέση κλειδί, είναι από τις πιο βασικές βιομηχανίες. Δεν μπορούμε λοιπόν να ε, τις επιβάλλουμε ουτοπικούς ανεδαφικούς στόχους, κάτι που θα βλάψει την, αποτελεσμα... την ανταγωνιστικότητά της, ε, θα προκαλέσει μεγάλο πλήγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία και θα μειώσει τις θέσεις απασχόλησης, χωρίς ταυτόχρονα να συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών. Και το 15% μέχρι το 2025 μείωση ήταν ε, εντάξει, αλλά δεν συμφωνώ με την φιλόδοξη ε, μείωση μέχρι το 2030 όπως προβλέπει η συμφωνία. Ευχαριστώ κύριος Μπουσόη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είδαμε ότι 500.000 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Οι πρωτεύουσε λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνουν ένα χειρομήνυμα. Θα πρέπει σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο να είμαστε φιλόδοξοι, χωρί να θέτουμε ένα αμφιβόλο, χωρί να υπονομεύουμε την αντιγωνιστικότητα τη αυτοκινητοβιομηχανία. Μετά τι θεσμικέ διαπραγματεύσει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να καταλήξει σε μια συμφωνία για την μείωση των εκπομπών κατά 37,5% για τα νέα οχήματα και 30% όσον αφορά τα επαγγελματικά οχήματα. Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά, λέει ο Πρόεδρος. Είμαι πεπισμένο, κύριε Πρόεδρε, ότι οι ποσοστώσει αυτέ που είναι ιδιαίτερα φιλόδοξε, τα ανώτατα αυτά όρια, θα πρημοδοτήσουν ακόμα περισσότερο την ανταγωνιστικότητα ανάμεσα στους κατασκευαστές αυτοκινήτων και θα καταφέρουμε να καταλήξουμε όντω σε οχήματα τα οποία έχουν πολύ χαμηλές ακόμα και μηδενικέ εκπομπές. Ευχαριστώ. Και τελευταίο ομιλητή στη διαδικασία Κατσδιάη, ο κύριο Δρογεύσκη. Ένα λεπτό. Δεν είναι σίγουρα η βέλτιστη λύση, είναι μια συμβιβαστική λύση. Απέχει από την ιδανική, γιατί με την ιδανική λύση, την βέλτιστη, όλοι είναι ικανοποιημένοι. Ενώ από το συμβιβασμό δεν είναι κανείς απόλυτα ικανοποιημένο. Οι οικολόγοι θα ήθελαν περισσότερες, πιο αυστηρές προδιαγραφές, πιο φιλόδοξους στόχους, ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία, οι χρήστες αυτοκινήτων μας επισημαίνουν το κόστος που θα έχει υπερβολικά γρήγορη και φιλόδοξη εφαρμογή των στόχων. Επίσης, μην ξεχνούμε την αυτοκινητοβιομηχανία και να μην μπερδεύουμε τους απλούς χρήστες ε, των ΙΟΤΑΧΗ με τους ε, επαγγελματίες. Επίσης, ε, πολλές φορές ο υπολογισμός του κόστους γίνεται ε, ξεχωριστά και κατακαιρματισμένα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς σωστά, ισορροπημένα και σταθμισμένα θα εφαρμόσουμε στην πράξη αυτές τις διατάξεις. Ευχαριστώ. και τώρα το λόγο έχει ο Επίτροπος, ο κύριος Αρίας Κάνιετ, εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε παρακαλώ να κάνετε μια σύνοψη κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση που δείχνει και πάλι τη μεγάλη σημασία τη σχετική νομοθετική πρόταση. Έχουμε και και τώρα ένα σχέδιο κλειδί για να εφαρμόσουμε το σχέδιο δράση για το περιβάλλον ανάπτυξη του 2030 και να εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις μας στη Συμφωνία των Παρισίων. Ο σχετικός κανονισμός δεν προστατεύει μόνο το περιβάλλον, αλλά θα βοηθήσει και τη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κρατήσει την πρωτοκαθεδρία της και την ανταγωνιστικότητά της σε μια ραγδαία μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά, όπου ε, η απέτηση επιχειρησιακών μοντέλων που στηρίζουν τη βιώσιμη κινητικότητα αυξάνεται. Επίσης, ε, με τα νέα μέτρα θα αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης, η κατανάλωση, οι επενδύσεις στις υποδομές, η μείωση των εισαγωγών και οι οικονομίες στον τομέα των συστοιχειών. Όλα αυτά είναι σημαντικά για να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Η σχετική νομοθεσία θα έχει πολλά οικονομικά ωφέλη και για τους καταναλωτές που δεν θα έχουν μόνο καθαρότερο αέρα, αλλά θα, θα εξοικονομήσουν χρήματα. Ε, και στα, στην κατανάλωση των οχημάτων τους. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε υπερήφανοι από το αποτέλεσμα των κοινών προσπαθειών μας. Γνωρίζουμε τι προσπάθειες θα χρειαστούν για να υλοποιήσουμε τις υποσχέσεις μας για το περιβάλλον και φάνηκε από τα συμπεράσματα της συζήτησης. Αυτός ο κανονισμός είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό παρακαλώ στην αυριανή ψηφοφορία να υπερψηφίσετε την έκθεση ώστε να τεθεί το νομοθέτημα αυτό το συντομότερο δυνατό σε ισχύ. Δεν έχουμε χρόνο να χάνουμε στον αγώνα μας κατά των κλιματικών αλλαγών γιατί περιμένουν από εμά οι πολίτες και σίγουρα και οι μελλοντικέ γενιές. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Ντάλη, η εισηγήτρια, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφου και να αναφερθώ σε κάποια από τα ζητήματα που εθίγησαν. Καταρχάς, α σταματήσει αυτό ο εκφοβισμός. Λέμε ότι οι περισσότερε επενδύσεις από τις επιχειρήσεις οδηγούν σε αυξανόμενο κόστος. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όλε οι έρευνε που έχουμε δει, ακόμα και εκτίμηση επιπτώσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν οικονομικά ωφέλη για του καταναλωτέ. Όπω το είπε τώρα μόλι ο ίδιο ο Επίτροπο, όταν αναφέρθηκε σε μείωση του κόστου για του καταναλωτέ. Το όφελο για του καταναλωτέ είναι, αν θέλετε, το πρώτο πράγμα το οποίο φαίνεται το θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την πρόταση κανονισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν ακριβώ τι λεπτομέρειε ε, οι συνάδελφοι που θα ψηφίσουν αύριο. Ο κ. Νότερ δεν κατάλαβε, για παράδειγμα, ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για αυτοκίνητα τα οποία εκπέμπουν 0,7% και ε, συνάδελφοι από το ECR δεν κατάλαβαν επίση ότι όλα αυτά αποτελούν ε, αναπόσπαστο τμήμα τη δέσμη μέτρων που έχουν να κάνουν με διάφορου τομεί ε, και ότι εμεί αυτή τη στιγμή δεν επικεντρωνόμαστε αναγκαστικά μόνο στην κινητικότητα ή στα επιβατικά αυτοκίνητα. Όντω οι αλλαγέ λαμβάνουν χώρα, έχουμε νέε επενδύσει σε νέε τεχνολογίε και διεξάγεται και έρευνα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί όντω να παράγει συσσωρευτέ και κυψέλε καυσίμου στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε χώρο επίπεδο και χαίρομαι πάρα πολύ που ορισμένοι συνάδελφοι που είχαν κάνει προτάσει λιγότερο φιλόδοξε στην αρχή, σήμερα φαίνεται να συμφωνούν και μιλάνε θετικά για τον συμβασμό που έχουμε ενώπιον μα. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι η αρχική φιλοδοξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν πραγματικά να αλλάξει τα πράγματα και να συνεχίσει να τροποποιεί τα πράγματα και στο μέλλον. Δείτε αυτή τη στιγμή τα διάφορα πρότυπα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται πλέον και δείτε επίση τα χιλιόμετρα τα οποία μπορούν πλέον και διανύουν τα οχήματα αυτά, τα οποία θεωρούνται οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών. Κάτι το οποίο δεν ίσχυε στο παρελθόν. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε την εργασία μας αυτή, α προσελκύσουμε περισσότερε επενδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ας δημιουργήσουμε την κατάλληλη υποδομή, τους κατάλληλους σταθμούς φόρτισης, καθώς επίσης και την απαραίτητη τεχνολογία προκειμένου να κατασκευάσουμε συσσωρευτές και κυψέλες καυσίμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Προσβλέπω στη θετική ψήφο σας αύριο. Ευχαριστώ και σας κύριε Επίτροπε και ευχαριστώ και το Σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξή της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν τη συζήτηση. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Η ψηφοφορία της έκθεσης Ντάλι θα λάβει χώρα αύριο. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα, στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που προβλέπει η συζήτηση της έκθεσης του κυρίου Παντσέρη και του κυρίου Πρέντα, του κυρίου Έγκελ και του κυρίου Γκέρενς με θέμα το Μηχανισμό γειτονία, Ανάπτυξης και διεθνού συνεργασία. Πρώτος λαμβάνει το λόγο ο ένας από τους συγγητές, ο κύριος Παντσέρη. Για τέσσερα λεπτά παρακαλώ. Μια στιγμή, μια στιγμή να προλάβει ο Επίτροπος να λάβει θέση και να βάλει τα ακουστικά του. Ευχαριστώ και σας ακούμε κύριε Παντζέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αύριο θα κληθούμε να υπερψηφίσουμε τη νέα αυτή θέσπιση μηχανισμού γειτονία, ανάπτυξη και διεθνού συνεργασία. Πρόκειται για μια διαδικασία πολύ σημαντική, γιατί θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο η υποστήριξη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προ τι τρίτε χώρε θα διευρυνθεί την περίοδο 2021-2027. Αναφερόμαστε λοιπόν εδώ πέρα περίπου σε 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κείμενο αυτό αποτελεί αποτέλεσμα μια μακρόχρονη συνεργασία και διαπραγμάτευση με όλε τι πολιτικέ ομάδε. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια τοποθέτηση που θεωρώ ότι είναι ισορροπημένη όσον αφορά τα διάφορα υφιστάμενα μέσα εξωτερική χρηματοδότηση, προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε έναν καλύτερο έλεγχο και επίβλεψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το τονίζω. Το ζήτημα τη διακυβέρνηση δηλαδή. Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μόνο εκτελεστικέ πράξει και συνέχιση τη επιτροπολογία για την έγκριση των κειμένων προγραμματισμού. Αυτό όμω σημαίνει στην πράξη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει πολύ περιορισμένη δράση στην περίπτωση αυτή. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε λοιπόν να εγκρίνουμε περισσότερε αποφάσει, ιδίω για τον προγραμματισμό όσον αφορά τι κατεξοδότηση πράξη. Μέσω των πράξεων αυτών μπορούμε να επέμβουμε πιο ουσιαστικά στο μηχανισμό αυτό και να επέμβουμε πραγματικά σε αποφάσει που λαμβάνονται για τον προγραμματισμό. Κατά αυτόν τον τρόπο, όλε οι σημαντικέ στρατηγικέ επιλογέ θα υπόκεινται στην εποπτεία και την παρακολούθηση αλλά και την ένσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Α μην ξεχνάμε ότι ε, η πολιτική γειτονία αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα για μα και αποτελεί, αν θέλετε, ένα έμβλημα τη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε μέσω του μηχανισμού αυτού να έχουμε την απαραίτητη ευελιξία, προκειμένου όντω να καταλήξουμε σε μια πολύ γρήγορη κινητοποίηση των επιπρόσθετων κονδυλίων που ενδεχομένω να απαιτηθούν για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Τα 92 δισεκατομμύρια αυτά τα οποία ανέφερα στην αρχή τη παρεμβασή μου, ουσιαστικά συνάδουν με τα κονδύλια τα οποία έχουν ήδη δεσμευτεί στα πλαίσια του νέου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου όσον αφορά την Αφρικανική Ήπειρο, εστιαζόμαστε στην υποσαχάρια Αφρική καθώ επίση και στι χώρε ΑΚΕ, ιδίω για να καλύψουμε το κενό το οποίο θα προκύψει μετά την λήξη τη υφιστάμενη συμφωνία Κοτονού η α, κατάργηση τη φτώχεια, η καταπολέμηση τη ένδυα, η πρόθεση τη αναπτυξιακή συνεργασία. Βλέπετε εδώ πέρα ότι προβλέπεται μία, ένα ποσοστό τη τάξη του 92% όσον αφορά τη χρησιμοποίηση τη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Χρειαζόμαστε επίση για τη μετανάστευση μια ολιστική προσέγγιση και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τα βαθύτερα αίτια της παράτυπης μετανάστευση, καθώς επίσης και των αναγκαστικών εκτοπισμών. Επίσης, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις κλιματικές αλλαγέ στα πλαίσια του μηχανισμού αυτού. Άρα, οι πολιτικές που θα εγκρίνουμε θα πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένε περιβαλλοντικές πολιτικές και επίσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίω όταν αναφερόμαστε στη μετανάστευση. Όσον αφορά τι κλιματικέ αλλαγέ, θα πρέπει εδώ πέρα να λάβουμε υπόψη μα τη Συμφωνία των Παρισίων και τι υπόλοιπε εγκριθήσει συμφωνίε και βλέπετε εδώ πέρα ότι υπήρξε μια αύξηση τη τάξη 45% όσον αφορά τη χρηματοδότηση για την μετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Ιδιαίτερα φιλόδοξη πρόταση αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να επέμβουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει μια ρήτρα αναστολή τη βοήθεια, αν δούμε ότι υπάρχουν συνεχεί παρατυπίε ή παραβίε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτε χώρε. Όσον αφορά το μέσο αυτό για την ειρήνη και τη σταθερότητα, θεωρούμε ότι οι πόροι για τον τομέα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να έχουμε πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη και σε καμία περίπτωση τα κονδύλια αυτά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά όπλων υπηρομαχικών ή για την προώθηση τη άμυνα ή των στρατιωτικών στόχων. Η έκθεση αυτή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική, μα απασχόλησε για πολλού μήνε και γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω και του τρει υπόλοιπου συνεισηγητέ για την πολύ κοινή επικοδομητική εργασία που είχαμε και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε την πρόταση αυτή. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Παντζέρη. Περάμε στου υπόλοιπους εισηγητές. Ο κύριος Πρέντε επίση για τέσσερα λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσοι παρακολούθησαν εκ του σύνεγγυ τη συζητήση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί τη προτάσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό, δεν θα εκπλαγούν που από του τέσσερι συνεισηγητέ, εγώ ήμουν εκείνο που είχε από την αρχή του περισσότερου ενδιασμού ω προ την ιδέα ενός ενιαίου μηχανισμού. Θα ήθελα λοιπόν να σα παραθέσω εν συντομία τι αιτίε αυτών των επιφυλάξεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και ένα χρόνο και περίπου είχε εκφράσει μια πολύ ξεκαθαρή θέση, ζητώντα ξεκάθαρα μέσα για την προεταξιακή διαδικασία, την ανάπτυξη, τη γειτονία και την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων ε, αυτών των πολιτικών αλλά και του οικονομικού σκέλου τέτοιων παρεμβάσεων. Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εξαίρεση τα προταξιακά μέσα δεν έλαβε είναι υπόψη την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατέθεσε την σημερινή πρόταση που συγχωνεύουν μια δεκαριά περίπου μηχανισμούς από προηγούμενα προγράμματα. Τον Ιανουάριο του 2018 το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα τάχθηκε κατά της ιδέας ενιαίου μηχανισμού για τις εξωτερικές δράσεις και δήλωσε απερίφραστα ότι αυτό αποτελεί ψευδέστηση απλούστευσης που θα οδηγούσε σε ατέρμονες εσωτερικές διενέξεις για το ποια βοήθεια είναι πιο σημαντική και ποιο μέσο είναι ο πιο σημαντικός. Το ΕΛΚ επισήμανε επίση ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική γειτονία που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών ε, με τη συγχώνευση αυτή θα υποσκαπτόταν και θα ε, χανόταν σε, χωρίς ένα δικό της ξεχωριστό χρηματοδοτικό μέσο. Παρόλα αυτά και παρά τους επιφυλάξεις μας, με υπεύθυνο τρόπο συμμετείχαμε στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να βελτιώσουμε την αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν ένα μακρόπνο έργο, δεδομένης της εξαιρετικής περιπλοκότητας του θέματος αυτού, που προϋποθέτει διάφορες ε, συζητήσεις και συμβασμό μεταξύ μερικές φορές και αντιφατικών ε, συμφερόντων και πρόκειται πραγματικά για επανάσταση σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η επανάσταση ανταποκρίνεται σε επανειλημμένα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μεγαλύτερη ελαστικότητα προκειμένου να ανταποκριθούμε σε απρόβλεπτες, απροσδόκητες προκλήσεις ε, σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση επίση και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είχαμε αρκετέ διευκρινήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε ξεκάθαρη, ε, και σαφή ορισμό των διαφόρων πολιτικών που καλύπτονται και των ε, οικονομικών εγγύσεων για την κατανομή των κονδύλιων και τη χρήση του. Χάρη στη συνεργασία πάντω των πολιτικών ομάδων, καταφέραμε τελικά να προτείνουμε ένα ισορροπημένο κείμενο για να εξασφαλίσουμε ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έλεγχό του, κυρίω χρησιμοποιώντα ε, τι κατεξουδότητε πράξει με ξεκάθαρου και φιλόδοξου στόχου για την εξωτερική δράση, θέτω στο επίκεντρο τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πρόθεση τη δημοκρατία, συνεννοηθήκαμε. Και σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά μέτρα, που είναι στο επίκεντρο τη συζήτηση, αυξήσαμε κατά 4,4% το συνολικό κονδύλιο του μηχανισμού, προσθέσαμε εγγυήσει για τι γεωγραφικέ οικονομικέ κατανομέ για την γειτονία και την υποστοχάρη Αφρική. Ενισχύσαμε τα κονδύλια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία των πολιτών και τις παγκόσμιες προκλήσεις, παράλληλα μειώνοντας ε, το αποθεματικό ε, από 10,2 σε 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας πόσο λυπάμαι για τη στάση των πρασίνων που στην ψηφοφορία στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ είχαμε δεχτεί πάνω από 250 δικές τους τροπολογίες, οι τέσσερις συνεισηγητές ε, συνολικά κατέθεσαν 380 τροπολογίες. Και παρά το γεγονός ότι δεχτήκαμε υπερβολικά μεγάλο αριθμό τροπολογιών ε, των πρασίνων, άνευ προηγουμένου κατάσταση για τέτοιου είδου έκθεση, παρόλα αυτά κρατήσατε στάση αποχή σε τελική ψηφοφορία. Προστή η συμπεριφορά. Ήταν ρεκόρ η αποδοχή των τροπολογιών σας και παρόλα αυτά θέλετε να χτυπήσετε το συγκεκριμένο μηχανισμό. Γιατί, θέλω απάντηση. Ε, τι θέλετε να κάνετε με αυτό το μηχανισμό και πώς αντιμετωπίζετε τη συγκεκριμένη ε, έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Έγγελ για τέσσερα επίσης λεπτά. Επίσης είναι εισηγητής maybe you, you can change the, αλλάξτε ε, θέση. Κύριε Πρόεδρε, να το θαύμα της τεχνολογίας συμβαίνει έστω και λίγο αργά σήμερα στην αίθουσα αυτή. Νομίζω ότι ξέρουμε για ποιο λόγο βρισκόμαστε εδώ πέρα και λυπάμαι. Λυπάμαι πραγματικά που είμαστε ελάχιστοι στην αίθουσα αυτή για μια δέσμη μέτρων η οποία αντιστοιχεί περίπου σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ για μια περίοδο προγραμματισμού 7 ετών. Αν θέλετε για ένα τέτοιο εγχείρημα θα περίμενα να ήταν λίγο περισσότεροι εδώ πέρα, αλλά ενδεχομένως η απουσία τόσο πολλών συναδέλφων να έχει να κάνει με το ότι ε, βρισκόμαστε πια στις τελευταίες εβδομάδες της κοινοβουλευτικής ε, θητείας. Όσον αφορά τώρα το κείμενο αυτό καθεαυτό, πρέπει να πω ότι Πρόκειται για ένα κείμενο το οποίο αντιστοιχεί πραγματικά στην αρχική φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν υπέβαλε την αρχική της ανακοίνωση. Όλοι όσοι εμείς που εμπλεκόμαστε στην, στην αναπτυξιακή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήρθαμε σε επαφή και με Αφρικανούς εταίρους οι οποίοι μας είπαν ότι υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης που μας προκαλούν πραγματικά σύγχυση. Ειλικρινά δεν ξέρουμε πού πρέπει να απευθυνθούμε προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη, πιο αποτελεσματική χρηματοδότηση. Ο ενίο λοιπόν αυτό μηχανισμό που θα θεσπιστεί θα επιφέρει και ένα υψηλότερο επίπεδο συνέπειας και συνεκτικότητος και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ θετικό χαρακτηριστικό. Αλλά κύριε Πρόεδρε, δυστυχώ υφίστανται ακόμα κάποιες αμφιβολίες, κάποιοι δισταγμοί γιατί ακόμα και αν υπερψηφίσουμε τελικά τη δέσμη αυτή μέτρων την οποία έχουμε προτιμάσει εμεί οι τέσσερι συνεισηγητές, αν συμβεί δηλαδή κάτι τέτοιο αύριο, θα πετύχουμε τον ευκταίο στόχο. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι ακόμα κρεμές. Το ζήτημα της συμπερίληψης του Ταμείου Ανάπτυξης στην, στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν πολιτικές ομάδες οι οποίες δεν θέλουν να ενταχθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης στο κοινοτικό προπολογισμό και αν τελικά δεν συμβεί κάτι τέτοιο δεν θα καταφέρουμε να έχουμε καθόλου ένα μηχανισμό γειτονίας ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας. Θα πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενισχύσει το μήνυμά του, που ήταν και το βασικό μήνυμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλωστε. Να καταφέρουμε να εντάξουμε στον κοινοτικό προπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη και θα πρέπει να συνταχθεί με τη θέση αυτή και το Συμβούλιο. Αντί αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο να βρίσκεται σε μια μεταπικιακή θα έλεγα στάση και να μην θέλει να εντάξει ενεργά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ε, στον κοινοτικό προπολογισμό. Και κρεμεί και ένα άλλο ζήτημα, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να ξέρουμε αν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όντως τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της πρότασης αυτής ή όχι. Διότι μου δίδεται η εντύπωση ότι όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες υπήρχε τουλάχιστον ένας επίτροπος και συνεργάτες του, ο οποίος προωθούσε όλο και περισσότερο την, το βασικό αυτό μέσο της πολιτικής γειτονίας και ότι θα έπρεπε ουσιαστικά επ' αυτού του μέσου να επικεντρωθούμε μόνο. Λες και η πολιτική γειτονίας αποτελεί τελικά αυτό σκοπό και από ό,τι φαίνεται, ο επίτροπο αυτό δεν θα μπορούσε να δεχθεί τη συμπερίληψη τη πολιτική γειτονία σε αυτό το νέο μηχανισμό. Α μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια επίσημη πολιτική τη Ένωση, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει απλώ με μια πρόταση του Συμβουλίου ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μιλάμε για 24% πρικοδότηση ουσιαστικά τη πολιτική γειτονία και από ό,τι φαίνεται και το ίδιο το γραφείο του Επιτρόπου για τη Διεύρυνση μας υπέβαλε κάποιες παρατηρήσεις κάποιες νουθεσίες που είχαν ως στόχο τελικά να ακυρώσουν όλη αυτή τη γενικότερη προσπάθεια θέσπισης ενός ενίου μηχανισμού. Θα μπορούσατε λοιπόν κύριε Επίτροπε να μου πείτε αν πραγματικά εξ αρχής τάχθηκε ομόφωνα της δέσμης αυτής μέτρων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή υπήρξε τελικά διάσπαση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την πρόταση αυτή. Του των λεχθέντων κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό συνεκτικό κείμενο και πραγματικά ελπίζω να υπερψηφίσετε αύριο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ και ο τελευταίο από του συνεισηγητέ, ο κύριο Γκέρεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω του συναδέλφου συνεισηγητέ, γιατί πιστεύω ότι επιτελέσαμε ένα πολύ αξιόλογο έργο το τελευταίο εξάμεινο και καθόλου εύκολο. Καταφέραμε παρόλα αυτά να σας υποβάλουμε μια έκθεση και πριν το πέρας της κοινοβουλευτικής μας Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους ε, της Επιτροπής Ανάπτυξης, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γιατί επέδειξαν ένα μεγάλο επαγγελματισμό, ανθεκτικότητα, αφοσίωση, επιμέλεια, ικανότητες καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των εντατικών προσπαθειών, γιατί είναι α, ίσως η πιο περίπλοκη έκθεση Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Μια άλλη καινοτομία ήταν ότι είχαμε συναρμοδιότητα τριών επιτροπών ε, που ασχολούνται με εξωτερικά θέματα. Ήταν λοιπόν ε, ρηψοκίνδυνο εγχείρημα. Και ήταν ρυψοκίνδυνο γιατί αναθέσαμε την έκθεση σε τέσσερις συνεισηγητές και τρεις επιτροπές. Ήταν επίσης ρηψοκίνδυνο το εγχείρημα αυτό, γιατί προσπαθήσαμε να ξεφύγουμε από την πεπατημένη χωρίς ταυτόχρονα να θυσιάσουμε τα κεκτημένα της ανάπτυξης. Ήταν ρηψοκίνδυνο επίσης το εγχείρημά μας, γιατί να καταφέρουμε μια σύγκληση απόψεων για το νέο αυτό μηχανισμό δεν ήταν κάτι δεδομένο ή αυτονόητο. Η κυρία Μογκερίνη είχε πει στην πρώτη παρουσίαση του εγγράφου που έκανε ότι οι πολιτικές θα διαφυλαχθούν ως προς την πεμπτουσία τους. Οι μέθοδοι όμως θα αλλάξουν. Και εμείς δεχτήκαμε αυτή την πρόκληση και δώσαμε έμφαση στην αλλαγή και τα καταφέραμε. Ξεφύγαμε λοιπόν από από την πεπατημένη για να καταστήσουμε πιο συνεκτικές τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βγήκαμε από την πεπατημένη προτείνοντας εγγραφή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό. Είπαμε λοιπόν να υπαχθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης στον κοινοτικό προϋπολογισμό, γιατί συνήθως ε, δίναμε κηρύγματα περί δημοκρατίας στον υπόλοιπο κόσμο, ενώ εμείς οι ίδιοι δεν είχαμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε μία ε, συναρμοδιότητα σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Επίσης, ε, βγήκαμε από την πεπατημένη και αντιληφθήκαμε ότι οι προκλήσεις αυτές ε, είναι άλλης κλίμακος για την περίοδο 2020-2027, πολύ διαφορετικές από τις τρέχουσες προκλήσεις. Επίσης, ε, βγήκαμε από την πεπατημένη και ε, παραδεχτήκαμε και ομολογήσαμε ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα, γιατί χρήματα λείπουν από παντού. Οπότε ήταν φυσιολογικό να καλέσουμε και τον ιδιωτικό κλάδο, τον ιδιωτικό τομέα να αφιερώσει ένα τμήμα των οικονομιών του και των μέσων του και των αποταμιεύσεών του στην ανάπτυξη. Και γι' αυτό με τη μόχλευση που θα δημιουργήσει ο ενιαίος μηχανισμός θα έχει περισσότερα μέσα να αφιερώσει από ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και τα κονδύλια της μόνο. Θα ήθελα να πω επίσης ότι ε, ενισχύονται και οι εξουσίες ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα θέματα αυτά, εφόσον η, ε, η Ολομέλεια εστερνιστεί τις προτάσεις μας και τις συστάσεις μας γιατί έγιναν σεβαστέ οι απόψει μα για θέματα διεθνού συνεργασία, έγιναν σεβαστέ οι εξουσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβάνοντα τις διάφορες απόψεις που υιοθετήσαμε τα τελευταία χρόνια για το θέμα αυτό και επίσης, και δεν είναι καθόλου ισονοσημασίας, έχουμε προηγηθεί του Συμβουλίου. Εμείς είμαστε έτοιμοι, γιατί αυτό ήταν το στίχημα, να ολοκληρώσουμε την ε, έκθεσή μας πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας και καταλήξαμε σε μια πολύ ισορροπημένη έκθεση για το μέλλον των εξωτερικών δράσεων της γειτονία και της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης και τα καταφέραμε. Ευχαριστώ. Τώρα, εκ μέρου τη Επιτροπή Προπολογισμών, το λόγο έχει η κυρία Γκορδία Σάμπαλ Ρουμπιάλ. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και η Επιτροπή Προπολογισμών προσπάθησε να ευθυγραμμίσει την πρόταση με την ε, θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Και από αυτήν την άποψη αυξήσαμε τα κονδύλια του νέου μηχανισμού ώστε να λάβει υπόψη και τις κλιματικές αλλαγές. Αυξήθηκε κατά 35% το σχετικό κονδύλιο και επίσης αυξήσαμε το κονδύλιο κατά 4 περίπου δισεκατομμύρια ε, σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις ε, για την Αφρική. Επίσης, μειώσαμε το μέγιστο ποσό του αποθεματικού στα 10 δις για να αποφύγουμε ανισορροπία μεταξύ των επιδοτήσεων και των χρηματοδοτικών μέσων και προβλέψαμε ένα μηχανισμό με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη χρήση του αποθεματικού που προβλέπεται στο Ταμείο αυτό. Επίσης, ε, ε, εγγυηθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ελάχιστο όγκο ε, επενδύσεων στο δημόσιο τομέα, ώστε να μην παρεμποδιστούν από τη μετάβαση στο νέο μηχανισμό. Και τέλος, ε, ε, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμη Ανάπτυξης και εκεί προσδιορίσαμε τον ορισμό της προσθετικότητα, Έχουμε πιο αυστηρά κριτήρια για την καταπολέμηση της ε, φορολογική απάτης, της λεύκασης του ξεπλήματο χρήματο και της κατάταξη τη φοροαποφυγή και βελτιώσαμε και το μηχανισμό υποβολή αιτιάσεων. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Επίτροπος Μίμητσα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους εισηγητές και όλους σας για την δουλειά που κάνατε στις Επιτροπές Εξωτερικών Προϋπολογισμού και Ανάπτυξης που οδήγησαν στην έγκαιρη ολοκλήρωση της έκθεσης ε, για την πρόταση αυτή. Χαίρομαι για το ότι η έκθεση στηρίζει συνολικά την φιλοδοξία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλωσορίζω ιδιαίτερο στην στήριξη του Κοινοβουλίου ένα πιο μέσο το οποίο θα είναι πιο συνεκτικό. Η φωνή της Ευρώπης στον κόσμο θα γίνει δυνατότερη και οι προτεραιότητες της θα εξυπηρετηθούν καλύτερα προτεραιότητες όπως η γειτονία, η υποσαχάρη Αφρική, η εξάλληψη της φτώχειας, η βιώσιμη ανάπτυξη, η μετανάστευση, η προώθηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, ε, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, διατήρηση της ειρήνης. Επίσης χαίρομαι που βλέπω ότι το Κοινοβούλιο διατήρησε τις επενδύσεις ως κάτι το οποίο θα πρέπει να κινητοποιηθεί για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους προσωπικά είμαι πεπισμένος για την ένταξη του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου στον ε, κοινοτικό προπολογισμό που θα ενισχύσει ιδιαίτερα τους ε, ελεγκτικούς ε, και δημοσιονομικούς ρόλους του Κοινοβουλίου. Όλα αυτά τα στοιχεία θα συνεισφέρουν στο ότι το νέο αυτό μέσο θα επιτύχει τους στόχους και τις δεσμεύσεις μας και την ε, παγκόσμια επίσης ατζέντα του 2030 στο πλαίσιο της συμπερίληψης ε, της ε, χρηματοδότησης του σκανδιναβικού μέσου που πρότεινε ομόφωνα η Κομισιόν θα ήθελα να τονίσω ξανά το εξής μια πιο αποτελεσματική αρχιτεκτονική των εξωτερικών δάπανών μας δεν αμφισβητεί την πολιτική σημασία οποιασδήποτε γεωγραφικής ή θεματικής πολιτικής αντιθέτως. Θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο της ε, κάθε πολιτικής με το να βελτιώνεται η ικανότητά μας για να κινητοποιήσουμε επιπλέον πόρους όπου αυτό απαιτείται. Αυτό είναι ιδιαίτερος ε, σημαντικό σε σχέση με απρόβλεπτες εξελίξεις, παραδείγματος χάρη στη γειτονιά μας. Στην ε, περιφέρειά μας ε, ο προγραμματισμός ακριβώς ε, θα μας οδηγήσει στην σύνθεση με την εφαρμογή των στόχων της χιλιετίας και των δικών μας συμφερόντων και των συμφερόντων των γειτόνων μας. Αυτό θα έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα μόνο εάν είναι ευέλικτο. Επίσης, καλωσορίζω την πολιτική φιλοδοξία Τη έκθεση να εστιάσει σε βασικές ε, προτεραιότητες όπως η ανθρώπινη ανάπτυξη ή η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Θεωρώ όμως ότι τέτοιοι στόχοι θα πρέπει να είναι φιλόδοξοι και όχι νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις. Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να περιοριστούν οι δραστηριότητε μα σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι περίπλοκο και μεταβάλλεται συνεχώ. Επαναλαμβάνω την πεποίθησή μου πώ. Οι φιλοδοξίες της ε, Κομισιόν αντικατοπτρίζονται πλήρως σε αυτήν την πρόταση και καλωσορίζω την στήριξή σας όμως στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030 ε, ένας ε, στόχος επίτευξης κατά 95% ίσως να μην είναι ρεαλιστικός. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε ένα σημαντικό βαθμό ευελιξίας όσον αφορά ακριβώς την ε, πρόληψη συγκρούσεων και την ειρήνη, τη συνεργασία με βιομηχανοποιημένες χώρες. Θεωρώ ότι με να ε, προτείνει η Κομισιόν ένα 92% ήδη είμαστε αρκετά φιλόδοξοι. Η Κομισιόν είναι έτοιμη να έρθει σε επαφή με το Κοινοβούλιο για να δούμε πώς θα μπορέσουμε καλύτερα να ενισχύσουμε τον ρόλο τον εποπτικό του Κοινοβουλίου. Ένα ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο είναι πράγματι ο στόχος μας. Σεβόμενη πλήρως την διοργανική ισορροπία. Όμως, θεωρώ ότι η δημιουργία επιπλέον στρωμάτων θεσμικού ελέγχου και η υπερβολική χρήση των πράξεων κατεξοδότηση δεν θα επιτύχει αυτόν τον στόχο. αυτού, θα καταστήσει την ε, λειτουργία του μέσου αυτού πολύ περιπλοκή. Έχει μεγάλη σημασία η επαρκής ε, φιλοδοξία. Στο πλαίσιο αυτό, το μέσο για την άμεση αντίδραση θα πρέπει να διατηρηθεί στον ε, ε, ε, κυβερνητικό πυλώνο. μαξιλάρι αυτό θα μας δίνει την απαιτούμενη δυνατότητα να αντιδρούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά σε απρόβλεπτες ανάγκες που είναι τόσο κοινέ στην εξωτερική δράση στην γειτονία και παραπέρα. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι τα αδιάθετα κονδύλια για το μαξιλάρι αυτό θα πρέπει να μειωθούν. Ούτε θα πρέπει να γίνει πιο περίπλοκη η κινητοποίησή τους. Αναμένω λοιπόν την συζήτηση και την αυριανή ψηφοφορία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Mr. Commissioner. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Η κυρία Σχάκ έχει το λόγο για ένα λεπτό εκ μέρους Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Λειτουργεί το μικρόφωνο. Τέλεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, χρειαζόμαστε μια πιο αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων και μεγαλύτερη λογοδοσία. Και γι' αυτό όταν η, πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη εξικέλευθε τροποποίηση ε, έδειξε ανοιχτό μυαλό. Πάντω, ο μόνο τρόπο για να αξιολογήσουμε κατά πόσο ο προτινόμενο νέο μηχανισμό που συγχωνεύει σε μία δημοσιονομική γραμμή πολλέ προηγουμένω ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι κατάλληλο προ το σκοπό που εξυπηρετεί και σωστή διαχείριση των κονδυλίων. Και αυτό είναι ακριβώ ακόμη τροτό σημείο στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταθέσαμε διάφορε προτάσει στην διευθύνουσα ομάδα μεταξύ της εξωτερικής δράσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σίγουρα η συνεργασία τους θα μπορούσε να έχει βελτιωθεί αλλά θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αιρεσιμότητα για τα δισεκατομμύρια αυτά ευρώ, μια πιο ελαστική εφαρμογή και φυσικά με τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με 1,6% μόνο του προπολογισμού να είναι αποθεματικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η δεύτερη μου προειδοποίηση είναι προ προσοχή να μην έχουμε εργαλειοποίηση της ε, εξωτερικής πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εντός εισαγωγικών διαχείριση της μετανάστευσης ή ε, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Και αυτό θα πρέπει να, φέρ, να φαίνεται και στον προπολογισμό για τις εξωτερικές υποθέσεις γιατί είναι σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού το λόγο έχει η κυρία Χιμένες Μπαρμπάτ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τις ε, τελευταίες δεκαετίες έγινε εμφανής η αύξηση των κοινών προκλήσεών μας. Γι' αυτό και το, ο νέο μηχανισμό γειτονία, ανάπτυξη και διεθνού συνεργασία είναι από τι πιο σημαντικέ προτάσει ε, τη τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία. Και αυτή η ρηξιγέλευτη αλλαγή στις, ε, στα μέσα εξωτερική ενίσχυση, τη εξωτερική χρηματοδότηση, θα ε, ενισχύσουν την ελαστικότητα και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο διεθνές προσκήνιο. Είναι σημαντικό λοιπόν οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από αυτό το μηχανισμό θα να συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, του θεματολογίου του 2030 και των Παγκόσμιων Συμφώνων. Και από αυτή την άποψη, στη γνωμοδότηση Επιτροπής ε, παιδείας και πολιτισμού δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τη σημασία της ποιοτικής χωρίς, περιορισμού, χωρίς Αποκλεισμού ε, παιδεία, που είναι σημαντικό κλειδί για να καταπολεμήσουμε την φτώχεια και τι ανισότητε και επίση ε, να τονώσουμε την ε, ανοχή να δημιουργώντας πιο φιλειρηνικές κοινωνίες και αντιμετωπίζοντας και τους βασικούς λόγους της μετανάστευσης. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίσουμε την χρηματοδότηση ευρωπαϊκής πολιτικής της γειτονίας και να ενισχύσουμε τη σύνδεση με τις χώρες της γειτονίας μας. Εκ μέρους τώρα της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το, υποσυζήτηση μηχανισμός είναι ένας, ένα γεωπολιτικό μέσο περισσότερο και όχι τόσο ένα μέσο ανάπτυξης. Λέμε ουσιαστικά ότι βοηθάμε τους μετανάστες ε, στις χώρες τους και ουσιαστικά οι προτεραιότητές μας έχουν να κάνουν με τα βασικά συμφέροντά μας στα πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής. Όλα γίνονται προκειμένου να σταματήσουν οι μεταναστευτικέ ροέ και να καταφέρουμε να περάσουμε από την παράτυπη μετανάστευση και παραθέτω εδώ πέρα την ίδια την έκθεση στην νόμιμη μετανάστευση. Α μην ξεχνάμε ότι η στάση μα αυτή τη στιγμή είναι ανεύθυνη πραγματικά. Κλασικά η πολιτική της ανάπτυξης ε, συνδυάζεται με την εξωτερική πολιτική και πολλές φορές ακόμα και με αμυντικούς και στρατιωτικούς στόχους. Και εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στρεφόμαστε κατά παλαιότερων ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ε, δεν λαμβάνουμε καθόλου υπόψη πολιτικές που έχουμε προωθήσει στο παρελθόν και που έχουν δημιουργήσει μόνο εξαθλίωση και ένδια. Α μην ξεχνάμε επίση ότι έχουμε πάρα πολλέ περιπτώσει καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα πρέπει το κακό να υπερτερεί σε πέντε στο καλό. Εκ μέρου τη Επιτροπή ε, Γυναικών και Ισότητα Ευκαιριών, η κυρία Φορέντζα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι συντάκτρια της γνωμοδότης Επιτροπής Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών όσον αφορά το νέο αυτό μηχανισμό Θεωρώ ότι είναι θετικό ότι ε, ασχοληθήκαμε στα πλαίσια αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου για το ζήτημα αυτό και ότι είχαμε και συνεργασία με πολλούς αρμόδιους φορείς. Πρέπει να σας πω πραγματικά ότι χρειάστηκε να αντιμετωπίσω ζητήματα ανάλογα με αυτά τα οποία ανέφερε πριν από λίγο και η συγγήτρια από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ουσιαστικά ένα κείμενο το οποίο θα έπρεπε να έχει ως στόχο να προωθήσει τι θεμελιώδει αρχέ ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ισότητα των φίλων ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντο και διαφορετικών πολιτισμών, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι ουσιαστικά γίνεται ένα κείμενο χρηματοδότηση συγκεκριμένων ταμείων και μέσων προκειμένου να καταφέρουμε να προστατεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μετανάστευση, προκειμένου να αναχαιτήσουμε το ίδιο το φαινόμενο τη μετανάστευση. Μολονότι έχουμε υποβάλει εμεί μια γνωμοδότηση ω Επιτροπή ΦΑΜ, πρέπει να πω ότι το τελικό κείμενο υπολείπεται όχι μόνο των στόχων τη Επιτροπή ΦΑΜ, αλλά ακόμα και το Gender Action Plan τη ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ζητήματα όπω τα δικαιώματα των γυναικών, η υποδέστερη θέση των γυναικών και βία κατά των γυναικών που δεν συμπεριλαμβάνουν στο διδακτικό του κειμένου, αλλά αναφέρονται σε καλύτερη περίπτωση μόνο στα παραρτήματα. Ο κύριο Μακάλιστερ το έχει το λόγο. Εκ μέρου του ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, να πω ω πρόεδρο τη ΑΦΕΤ ότι πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω του τέσσερι ηγητές για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν ο στόχος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελπίζω να είναι σαφής. Ε, πρέπει να φροντίσουμε η εξωτερική μας δράση να έχει επαρκή κονδύλια για να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση των αξιών μας παγκοσμίω. Η ευρωπαϊκή εξωτερική δράση πρέπει να είναι συνεκτική και ευέλικτη, δηλαδή να συγχωνεύει τα διάφορα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε ένα θεμελιώδες συμφέρον να ισορροπήσουμε την συνοχή με την δημοκρατική λογοδοσία. Οπότε ορίζω το ότι η έκθεση αυτή προβλέπει έναν ενισχυμένο διάλογο μεταξύ του Κοινοβουλίου μας και της ε, Κομισιόν και την χρήση των πράξεων κατεξουσιοδότηση για τις σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Νόιζερ, για δύο λεπτά από τους σοσιαλδημοκράτες. 100 δισεκατομμύρια ευρώ για 7 χρόνια. Ένα πολύ μεγάλο μέσο, το οποίο πολλοί συνάδελφοι βλέπουν με μεγάλη επιφύλαξη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους συζητητές και τους συναδέλφους ε, σοσιαλδημοκράτες όπως ο Αντώνιο Παντσέρη με τον οποίο συνεργάστηκα στενά. Θεωρώ ότι είναι μια πρόταση καλή, ένα ολοκληρωμένο πακέτο το οποίο αποφασίσαμε από κοινού να και στην ΔΕΒΕ. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια επιλεγμένα σημεία από την σκοπιά της αναπτυξιακής συνεργασίας καταφέραμε 45% αντί για 25% των μέσων αυτών θα πάει στο κλίμα, στην προστασία του περιβάλλοντος, ε, της βιοπικιλότητας και την καταπολέμηση της απερίμωσης. Δεύτερον, πετύχαμε να λαμβάνετε υπόψη σοβαρότερη μετανάστευση ως διεθνής πρόκληση και είναι σημαντικό ακριβώς η πολιτική αυτή να φροντίζει για την ασφάλεια των ανθρώπων όπως ακριβώς καθορίζεται στο διεθνές δίκαιο και στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μετανάστευση είναι απλά το επακόλουθο των συγκρούσεων της φτώχειας και θέλουμε ακριβώς να καταπολεμήσουμε τις αιτίες. Γι' αυτό 10% για την ε, μετανάστευση επίσης είναι πολύ σημαντικά. Θεωρώ ότι εμείς ως σοσιαλδημοκράτες ειδικά ε, πρέπει να χαιρετήσουμε αυτό το μέσο. Μιλάμε επίσης για την ισότητα των φύλων, συμμετοχή κοριτσιών και γυναικών. Είμαι πεπισμένος ότι είναι μια καλή βάση το μέσο αυτό και τα όσα ακούμε από την κοινωνία των πολιτών είναι πάρα πολύ θετικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ε, επικοδομητική συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Απ' την άλλη... Ε... 1,5 λεπτό η κυρία Βέχκα Περά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Μηχανισμός Γειτονίας Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας είναι μια πολύ φιλόδοξη μεταρρύθμιση της ε, εξωτερικής χρηματοδότησης, των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης και των εξωτερικών δράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υλοποιήσουμε και τους στόχους του θεματολογίου του 2030 και τους, βιο, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αν δεν τα καταφέρουμε θα σημειώσουμε παταγώδη αποτυχία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε μεγαλύτερη φιλοδοξία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε 45% της χρηματοδότησης να αφιερωθεί σε περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις. Επίσης, ε, συμπεριλάβαμε στο μηχανισμό την ανάγκη ενίσχυση της ισότητας των φύλων και στήριξη των προσπαθειών ε, ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της παιδείας και της υγείας. Τώρα που το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο ενεγράφει στον κοινοτικό προπολογισμό κάτι που ενισχύει το δημοκρατικό έλεγχο τη αναπτυξιακή βοήθεια, ελπίζω να συμφωνήσει και το Συμβούλιο και να εγκρίνει την υπαγωγή του ΦΕΔ στον προπολογισμό. Επίση, ενισχύουμε το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίω ό,τι αφορά τα μέσα εξωτερική χρηματοδότηση και την χρηματοδότηση των εξωτερικών δράσεων. Επίσης έχουμε τη συνεργασία μεταξύ της ε, βόρειας διάστασης και της ακτικής περιοχής, ε, βιώσιμη ανάπτυξη, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, ισότητα φύλων και εξάλληψη της φτώχειας. Ε, όλα αυτά ήταν, είναι και θα είναι εξαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές για τις εξωτερικές μας σχέσεις. Δεν αρκούν όμως μόνο οι στόχοι. Θα πρέπει να υλοποιούνται και εμπράκτος αυτοί. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό, εκ μέρου των Πρασίνων, το λόγο έχει ο κύριο Ρεϊμόν. Ευχαριστήσω τον Επίτροπο. Εμείς οι πράσινοι ήμασταν πάρα πολύ επιφυλακτικοί με το μέσο αυτό που συνενώνει τόσα πολλά χρηματοδοτικά μέσα προσπαθήσαμε να είμαστε επικοδομητικοί το πήραν πάρα πολύ σοβαρά όπως το είπε και ο κύριος Πέντα 200 ε, τροπολογίες ε, προσπαθήσαμε να κάνουμε πάρα πολλά. Ε, καταφέραμε κάποια πράγματα, κάποιοι εισηγητές πράγματι οδήγησαν σε μια επικοδομητική διαπραγμάτευση ποσοτικά έγιναν πάρα πολλά. Με την ποιότητα δεν είμαστε τόσο ικανοποιημένοι. Πάρα πολλά πράγματα στον τομέα προστασία του κλίματο, ισότητα των γυναικών, αλλά τα σημαντικότερα ζητήματα ε, κανονίζονται τελικά στα εκτιμώντας και τις παρατηρήσεις και όχι στο διατακτικό. Εμείς θέλαμε να διαπραγματευτούμε ακόμη περισσότερο και είμαστε διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουμε και τις τελευταίες στιγμές για να κάνουμε κάποια αποφασιστικά βήματα έτσι ώστε να δοθεί ακριβώς αυτή η τελευταία αλλαγή που θα μας επέτρεπε να υπερψηφίσουμε. Όπως είναι το κείμενο. Θα μπορούσαμε να ασκήσουμε σωστή πολιτική, αλλά δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση. Στον τομέα της μετανάστευσης θα μπορούσαν τα λεφτά να χρησιμοποιηθούν ε, σωστά, ε, οπωσδήποτε δεν θα το στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σάντζες Καλτεντέη, εκ μέρου τη ΓΚΟΑ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενοποίηση όλων των χρηματοδοτικών μέσων της εξωτερικής δράσης είναι προσβολή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί αγνοήσατε πλήρω το ψήφισμα τη 14η Μαου του 2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκεί που είχαμε ζητήσει συγκεκριμένα και ξεχωριστά μέσα και μηχανισμού για την διεθνή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια. Γι' αυτό απορρίπτουμε πλήρω την νομοθετική σα πρόταση, γιατί η συγχώνευση των ε, υπαρχών των ταμείων δεν σέβεται την βιώσιμη και την αναπτυξιακή πολιτική. Το αντίθετο κάνει, γιατί θα χρησιμοποιήσει τα αναπτυξιακά κονδύλια για να εξυπηρετήσει γεωστρατηγικά και αμυντικά συμφέροντα. Ο πραγματικό στόχο που κρύβεται πίσω από αυτή τη συγχώνευση των μέσων είναι η χρήση των αναπτυξιακών κονδυλίων για τον έλεγχο τη μετανάστευση, τον έλεγχο των συνόρων και για αμυντικού στόχου. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι πολίτε να ενημερωθούν ότι με την πρόταση αυτή θα σταματήσουμε να είμαστε ο πρώτο ε, δωρητή αναπτυξιακή βοήθεια στον κόσμο, κάτι που μα έκανε υπερήφανο. Από εδώ και πέρα τα κονδύλια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για. Ε, για περιπολίες στα σύνορα, για όπλα, για φράχτες και σειρματοπλέγματα. Ε, Απ' τη μια καταπατούμε τα ιδεώδη μας και απ' την άλλη ε, διαρωτόμαστε προς τι απογοήτευση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Τέτοιου είδους προτάσεις μας απομακρύνουν από τους στόχους μας και από τις διεθνείς μας υποχρεώσεις, όπως η ατζέντα για το 2030 ε, που συνεχώς ε, την αναφέρουμε, αλλά μόνο στα λόγια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλαφράνκα Σάτσε Νέιρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, κυρίε και κύριοι. Συνήθω ξεκινώ με συγχαρητήρια προ του συζητητέ για το έργο του. Αυτή τη φορά δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν συμφώνησαν οι δύο συνεισηγητέ τη ομάδα. Αλλά εδώ θέλουμε μια εξωτερική πολιτική πιο συνεκτική, πιο προβεβλημένη και πιο αποτελεσματική. Και αυτό το στόχο θα πρέπει να εξυπηρετούν τα δαψιλά κονδύλια του ενιαίου μηχανισμού. Νομίζω όμως ότι θα κάναμε λάθος συζήτηση αν τώρα συζητούσαμε αν πρόκειται για ένα ενιαίο μηχανισμό ή διαφοροποιημένο όργανο. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε βαρύτητα στο διεθνές προσκήνιο, ανάλογο με το βιομηχανικό, οικονομικό και πολιτικό μας δυναμικό. Θέλουμε μια συνεκτική πολιτική που θα προσαρμόζει τις μεταβαλλόμενες αλλαγές και προκλήσεις. Η ε, κυρία Σχάκη έφυγε από την αίθουσα. Αλλά, όπως είπε, σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, δεν πρέπει να κάνουμε λάθο συζήτηση. Το θέμα δεν είναι ενιαίος μηχανισμός ή διαφοροποιημένοι μηχανισμοί. Το θέμα είναι να δώσουμε έμφαση στην εξωτερική πολιτική και να προβάλλουμε την εξωτερική πολιτική και τι εξωτερικέ δράσει Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακάβαν για ένα λεπτό. Um, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία ήδη ακούστηκαν από τους συγητές και τους ομιλητές της ομάδας μου για τις τροπολογίες κλειδιά. Νομίζω ότι βελτιώνουν το κείμενο και ελπίζω να τις δεχτεί το Συμβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές, ειδικά τους κυρίους Έγγελ και Γκέρενς γιατί υπερασπίστηκαν την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική και θεώρησαν ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Βασίζεται στις αξίες, στην καταπολέμηση της φτώχειας και τον αγώνα για παγκόσμια δικαιοσύνη. Δύο πράγματα. Πρώτον, στην περίοδο που θα λειτουργήσει το μέσο αυτό, από τώρα μέχρι το 2030. Μιλάμε για μια κρίσιμη περίοδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιτύχει τους στόχους των Παρισίων και της ε, χιλιετίες για εμάς και για ολόκληρο τον πλανήτη. Και βεβαίως ε, θα αποτελέσει τμήμα της όλης διαδικασίας ε, η διαδικασία αυτή. Και μετά από 21 χρόνια, μάλλον τελευταία φορά που μιλάω ως Ευρωβουλευτής εδώ μέσα, να σας ευχαριστήσω λοιπόν κύριε Επίτροπε, σας και το προσωπικό σας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή ΔΕΒΕ και τους συναδέλφους ε, της ΑΦΕΤ και το προσωπικό και τους ευρωβουλευτές. Θα ήθελα να αναφέρω δύο άτομα όμως ε, ιδιαίτερα. Τους δύο βοηθούς μου στα θεωρία μου είπαν ότι απόψε είναι η πρώτη φορά που είχαν χρόνο να έρθουν γιατί εργάζονται. Οπότε να ευχαριστήσω τις ε, κυρίες Κέρι και ο Κόνορ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα κυρία Σαρχεντίνη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα έχουμε μια ατυχή κατασκευή. Η αναπτυξιακή πολιτική και η εξωτερική πολιτική δεν είναι πάντα το ίδιο. Η εξωτερική πολιτική συχνά είναι βράχη πρόθεσμη και φροντίζει τα δικά μας συμφέροντα, ενώ ε, η αναπτυξιακή πολιτική έχει στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας. Αυτά λέει η συνθήκη, καταπολέμηση της φτώχειας. Η συγχώνευση των δύο δημιουργεί τον κίνδυνο να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Και όταν λέει ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θέλει να εξοικονομήσει λεφτά για ευελιξία, τότε αρχίζω να ανησυχώ. Η αναπτυξιακή συνεργασία δεν έχει καμία δουλειά με την ευελιξία. Πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και προβλέψιμη. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι εμείς οι πράσινοι και δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι το σχέδιο Β εάν δεν επιτύχει αυτό. Γιατί βεβαίω δεν υπάρχουν και τα απαραίτητα λεφτά. Επίση, ε, η βραχυπρόθεσμη σκέψη δεν είναι κατάλληλη για την κλιματική πολιτική. Χαιρόμαστε ότι υπάρχει εδώ πέρα μία πρόταση για το 45% που πρέπει να πάει σε μέτρα του κλίματος. Προσπαθήσαμε να είμαστε πάρα πολύ επικοδομητικοί στις ε, προτάσεις μας. Χαιρόμαστε για το ότι έγιναν δεκτές οι προτάσεις μας, αλλά βεβαίω το θέμα εδώ είναι το αποτέλεσμα. Οι πράσινοι ε, συνεργάστηκαν σκληρά, αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις έτσι ώστε ε, να βλέπουμε κάποια ελπίδα για το ότι θα βοηθήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Κομισιόν στην καταπολέμηση της στόχης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Είναι μια τάση εδώ πέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει τα λεφτά που πήγαιναν για αναπτυξιακή βοήθεια και τα διαθέτει για άμυνα και ε, μετανάστευση. Το ίδιο και με το μέσο σταθερότητας και ειρήνης, με το καταπίστευμα για την Αφρική και τώρα με την ε, συνένωση αυτών των δύο ταμείων. Δηλαδή, ο στρατός ως αναπτυξιακή βοήθεια. Περιέχονται αυτά στην πρόταση της ε, Κομισιόν και προβλέπονται έτσι και από την Επιτροπή. Με τον στρατό σε περιοχές κρίσης δεν περιορίζεται η φτώχεια. Έχουμε το οριστικό τέλος μιας ουδέτερης ευρωπαϊκής πολιτικής βοήθειας σε περίοδους ε, κρίσης. Έχουμε λοιπόν μια συγχώνευση των ε, μέσων εις βάρος της ε, διαφάνειας και του δημοκρατικού ελέγχου. Έχουμε λοιπόν την συγχώνευσή τους πλέον και την αναπτυξιακή συνεργασία και υπάγονται όλα πλέον στην εξωτερική πολιτική και στα γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. Η συμπερίληψη μάλιστα στρατιωτικών επιχειρήσεων και των λεγόμενων ε, στρατιωτικών εταίρων ως ένα είδος μεταβατικής διοίκησης, δηλαδή ο στρατό